Let's start again. Last half session before the summer break. Λοιπόν, άντε, να τελειώνουμε αγαπητοί συνάδελφοι. And uh, hopefully there will be some further Λοιπόν, ξεκινάμε εμείς και ελπίζω να έρθει και κάποιος βουλευτής σιγά σιγά. Οι πολιτικές ομάδες, δεν ξέρω, έχουν ακούσει τίποτα, μήπως έρθει κανένας βουλευτής, ε, έχετε εσεί καμία ένδειξη. no, you are here. Yeah, yeah, yeah. So, because I think on item 14 Λοιπόν, επειδή το σημείο 14 είναι σημαντικό, ανταλλαγή απόψεων ε, με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ε, καλωσορίζω και πάλι την κυρία Κορίν Βάργα. Καλώς ήρθατε. Βεβαίω πάντα έχουμε αυτήν την συζήτηση όταν μιλάμε για εμπορικές συμφωνίες, για τι συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ως όρο και προϋπόθεση για να έχουμε δίκαιες εμπορικές συμφωνίες. Είχαμε φέτος την Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας 28 Μαΐου με 8 Ιουνίου και αναφέρθηκαν νομίζω οι περιπτώσεις 23 χωρών. Οπότε με τις οποίες θα έχουμε με τις οποίες έχουμε εμπορικές ε, συμφωνίες και έχουμε τις 8 βασικές ε, συμβάσεις ε, του ILO και βλέπουμε πως η Ιαπωνία δεν έχει κυρώσει την 105 και την 111 περί καταναγκαστικής εργασίας και διακριτικής μεταχείρισης και ο διάλογος ε, με τις Ιαπωνικές αρχές κατέστησε σαφές ότι χρειαζόμαστε μια δέσμευση για να σημειωθεί κάποια πρόοδος. Με το Βιετνάμ και την Σιγκαπούρη επίσης τρεις συμβάσεις ε, του ΑΙΛΟ δεν έχουν κυρωθεί. Βεβαίω δεν είναι εύκολο να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα εγκρίνει μια συμφωνία με έλλειψη σε αυτά τα σημεία. Οπότε η ανταλλαγή αυτή και η, συζή, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κυρία Βεργά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Είμαι η Κορίν Βαργά, Διευθύντρια του Τμήματος ε, Διεθνών Προδιαγραφών Εργασίας ε, στα κεντρικά μας στη Γενέβη. Το τμήμα το οποίο έχει δουλειά να λειτουργεί σωστά το εποπτικό σύστημα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, μόλις τελειώσαμε ακριβώς ε, την ε, διεθνή μας διάσκεψη ε, και συζητήσαμε 24 συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρών. Και με χαρά σας ενημερώνω ότι φέτος η Επιτροπή μας είχε πολύ καλές επαφές και συζητήσεις με τις ε, χώρες αυτές για τις οποίες υπήρχε η συζήτηση για την συμμόρφωση με τις σχετικές προδιαγραφές Να σας πω λοιπόν το εξής. Ζητήθηκαν 7 αποστολές από την Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προδιαγραφών, μια αποστολή ψηλοπέδου στην Αλγερία και 6 επαφές, έξι αποστολές άμεσων επαφών όπως τις λέμε, που θα γίνουν σε 6 έξι χώρες. Μπαχρέιν, Βολιβία, Ονδούρα, Μαλαισία, Μιανμάρ και Νιγηρία. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, προτείνω να σας ε, δώσω κάποιες ε, πληροφορίες για χώρες που μάλλον θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο και βεβαίως είμαι και στην διάθεσή σας μετά για ερωτήσεις ε, και απαντήσεις. Και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Όπως είπατε, ας ξεκινήσουμε με την Ιαπωνία την οποία αναφέρατε η Ιαπωνία είχε έρθει στην επιτροπή μας όσον αφορά την σεβασμή τη ΣΥΜΕΣ 87 για τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Ε, είχε κυρώσει την 65, το είχαμε συζητήσει 6 φορές στην επιτροπή μας ε, πέρσι και από το 2008. Τα ζητήματα αυτά που είναι αντικείμενο των συζητήσεων μη συμμόρφωσης αφορούν την άρνηση του δικαιώματος συνδικαλισμού στους δημοσίους υπαλλήλους, στους πυροσβέστες ε, και στους δεσμοφύλακες. Και υπάρχουν και κάποια ζητήματα που έθεσαν τα συνδικάτα όσον αφορά τις διαδικασίες αποζημίωσης ε, των εργαζομένων που δεν έχουν δικαίωμα απεργίας. Στις συζητήσεις ενώπιον της Επιτροπής η Ιαπωνία ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι είχε κάνει μια έρευνα τον Ιανουάριο που μας πέρασε για να δει τα προβλήματα που σχετίζονται με την λειτουργία του Συνδικάτου των Πυροσβεστών που επίσης απαγορεύεται να συνδικαλίζονται με σκοπό να βελτιωθεί η λειτουργία και αυτό έγινε σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους ε, η ΔΕ Επιτροπή για την Εφαρμογή των Πρωτογραφών σημείωσε με ανησυχία ότι τα ζητήματα αυτά είχαν τεθεί από την Επιτροπή των Ειδικών εδώ και δεκαετίες και τα προβλήματα παραμένουν. Οπότε στα συμπεράσματά τους ε, ζήτησαν ε, κάποιες συγκεκριμένες δράσεις που έπρεπε να αναλάβει η κυβέρνηση της Ιαπωνίας και πιο συγκεκριμένα ζήτησαν από την κυβέρνηση να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης με χρονοδιάγραμμα που θα εφαρμοστεί μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους για να εφαρμοστούν αυτές οι δεσμεύσεις ε, και οι συστάσεις της Επιτροπής και θα πρέπει να υποβληθεί πριν από τον Νοέμβριο φέτος στην Επιτροπή των Ειδικών για όσους δεν το γνωρίζουν. Η Επιτροπή των Ειδικών αποτελείται από 20 ανεξάρτητους ειδικού που δεν είναι προσωπικό του ΑΕΛΟ και συνεδριάζουν κάθε χρόνο στην Γενέβη και αφορούν ακριβώς την εφαρμογή των συμφωνημένων προδιαγραφών. Η κυβέρνηση λοιπόν στην απάντησή της επανέλαβε την δέσμευσή της για το ότι θα συνεχίσει να εξετάζει το τι θα γίνει στο μέλλον σε σχέση με τα ζητήματα αυτά που έχει θέσει το εποπτικό σύστημα εδώ και καιρό, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα, το εξή Ότι πριν ε, να είναι σε θέση να αλλάξουν την νομοθεσία θα χρειαστούν κάποια στήριξη από τους Ιάπωνες πολίτες και ε, για την ώρα δεν έβλεπαν ε, κάτι τέτοιο για αυτές τις αλλαγές. Οπότε συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας με την κυβέρνηση όπως κάναμε εδώ και καιρό. Τώρα, λίγα λόγια σε σχέση με το Μεξικό. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτή η χώρα σας ενδιαφέρει. Το Μεξικό ήρθε στην Επιτροπή σε σχέση με την Σύμβαση 87. Και πάλι δικαίωμα του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε και τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Ήδη είχε εμφανιστεί τρεις φορές ε, στην Επιτροπή μας. Τελευταία φορά ήταν το 2016, πρόσφατα λοιπόν τα ζητήματα της ε, μη ε, συμμόρφωσης βεβαίως ε, αφορούν και πράξεις βίασης βάρος των συνδικαλιστών μεταξύ των οποίων και δολοφονίες. Τα ζητήματα κάποιων παράτυπων συμβάσεων και ζητήματα που αφορούν τον πλουραλισμό στα συνδικάτα και την δυνατότητα να εκλέγουν επικεφαλής των συνδικάτων τους. Η Επιτροπή για την εφαρμογή των προδιαγραφών ε, ζήτησε περαιτέρω νομοθετική δράση και συνταγματική και όσον αφορά την ε, νομοθεσία και πάλι μέχρι τον ε, Νοέμβριο όπως ανέφερα είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή και με το Γραφείο και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ε, κυβέρνηση του Μεξικού για να προχωρήσει αυτές τις πολύ αναμενόμενες αλλαγέ. Σε δύο λόγια για την Μιανμάρ. Και η Μιανμάρ ε, ήρθε στην Επιτροπή μας ε, όσον αφορά τη Σύμβαση 87 πάλι, την οποία είχε κυρώσει το 1955. 18 φορές είχε έρθει στην Επιτροπή μας ε, από το 1987, τελευταία φορά το 2011. Οπότε είναι μια ιστορία που τραβάει εδώ και καιρό μεταξύ της ε, κυβέρνησης της Μιανμάρ και των εποπτικών φορέων ε, του ΑΕΛΟ και το ξέρετε αυτό φαντάζομαι. Το βασικό ζήτημα μη συμμόρφωσης ε, αφορά πάλι αστικές ελευθερίες, το δικαίωμα της ειρηνικής συγκέντρωσης και διαδήλωσης που έχει σοβαρότατους περιορισμούς η διαδικασία αυτή, την οποία γνωρίζω ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, έχει αποτελέσματα πάρα πολύ αργά και κάποια ζητήματα ακόμα πρέπει να αντιμετωπιστούν νομοθετικά και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ανησυχίες σε σχέση με τις ειδικέ οικονομικές ζώνες. Ε, για την ώρα δεν υπάρχει εγγύηση του δικαιώματος ε, του συνεταιρίζεστε στους εργαζόμενους ε, στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Και εδώ πέρα πάλι η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της ε, και την θλίψη της για το ότι δεν έχει υπάρξει κάποια πραγματική πρόοδος στο να εφαρμοστεί η νομοθεσία στις διάφορες διατάξεις που έχουμε τονίσει και ζήτησε μια αποστολή άμεσης επαφής για να πάει στη χώρα πριν από τον Ιούνιο του επόμενου έτους και να αναφέρει πάλι φέτος η χώρα στην Επιτροπή Ειδικών. Επίσης, τα περιθώρια της συνέλευσης ήμασταν σε επαφή με την κυβέρνηση για να προετοιμαστεί αυτή η αποστολή. Η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει η συνεργασία της και αναγνώρισε και ευχαρίστησε δημοσίως τις κυβερνήσεις μεταξύ των οποίων και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ε, και την Κομισιόν για την στήριξη που δίνουν στη Μιανμάρ και εξέφρασε την επιθυμία της να συνεργαστεί στενά με όλους και με τον οργανισμό μας για να προχωρήσει τα ζητήματα εργατικού δικαίου. Περνάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, την Γεωργία ε, η οποία μας απασχόλησε με την σύμβαση 100 που κύρωσε το 1993 δεν είχε έρθει ποτέ ενώπιον της Επιτροπής μας ε, έχουμε εδώ πέρα ζητήματα ίσης πληρωμής δεν υπάρχει νομοθεσία για την εφαρμογή της αρχής της ίσης πληρωμής για ίση εργασία και υπάρχει και ο νόμος ε, περί δημοσίων υπηρεσιών που ερμηνεύει στενότερα την ίση αμοιβή για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το, η κυβέρνηση ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είχε ένα εθνικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ε, μη διακριτικής μεταχείρισης ε, και της ίσης πληρωμής. Ταυτόχρονα αναγνώρισε ότι πρέπει να κλείσουν κάποια νομοθετικά κενά τα οποία εξετάζει και επίσης αναγνώρισε ότι οι επιθεωρητές, η επιθεώρηση εργασίας κυρίως ασχολείται με ζητήματα ασφαλείας και υγιεινής και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα υπόλοιπα και η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προδιαγραφών ζήτησε από την χώρα να κοιτάξει τα μέτρα επιβολής και μηχανισμούς ανείχνευσης που θα επέτρεπαν στην χώρα να επανορθώσει γρήγορα, καθώς το τωρινό μισθολογικό χάσμα είναι πολύ μεγάλο, για να δω, ναι. Το συνολικό χάσμα των φύλων στους μισθούς είναι 36%, πολύ σοβαρό, και το γνωρίζει αυτό η κυβέρνηση και η Επιτροπή ζήτησε από την χώρα να δώσει τεχνική αρρωγή και να επανέλθει τον Νοέμβριο για την τεχνική αρρωγή. Δύο λόγια. Να τονίσω εδώ ότι ένα από αυτά που προσπαθεί να κάνει το Διεθνής, Διεθνές Γραφείο Εργασίας είναι να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο ανάμεσα ε, στο εποπτικό σύστημα και το, την τεχνική αρρωγή. Όταν ε, προκύπτει πρόβλημα μη συμμόρφωσης, ε, ε, το οποίο εντοπίζει το υποπτικό σύστημα, αμέσως το γραφείο αναλαμβάνει να προσφέρει στη κυβέρνηση ροχή, στήριξη, βέβαια αν έχει δείξει ενδιαφέρον, και Έχουμε δει υποσχόμενα αποτελέσματα από την πρόθεση αυτού του νάρτου κύκλου ανάμεσα στην εποπτεία της εφαρμογής των υποχρεώσεων των κρατών μελών και την κατά προτεραιότητα παροχή τεχνικής αρρωγής. Και θέλω ταυτόχρονα να ευχαριστήσω την Trade και την DigiDevco της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους οποίους ε, συνεργαζόμαστε για στοχοθετημένη ε, τεχνική αρρωγή για να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη-μέλη που το χρειάζονται. Δύο λόγοι για τη Μολδόβα και την Ουκρανία. Ε, επιθεώρηση εργασίας εδώ ε, οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων έχει εκφράσει ανησυχία για το περιορισμένο πεδίο παρέμβασης των ε, επιθεωρήσεων εργασίας στις δύο χώρες. Πρέπει να ενημερώσουν προηγούμενα πριν να μπορέσουν να κάνουν οποιαδήποτε επιθεώρηση. Επίσης υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων και έχουν παρόμοια ζητήματα αποκεντρωμένων αρμοδιοτήτων επιθεώρησης σε τοπικό επίπεδο με απουσία σωστού συντονισμού. Και στις δύο λοιπόν περιπτώσεις η Επιτροπή Εφαρμογής των Προτύπων έχει ζητήσει από τις δύο χώρες να συνεχίσουν να ζητούν τεχνική αρρωγή ε, και Επίσης, είχε καλέσει τις δύο χώρες να αναφέρουν τι έχουν κάνει ενώπιον της Επιτροπής των Επιρογνωμόνων πριν το Νοέμβριο. Τώρα, εδώ και αρκετό καιρό ε, προσπαθούμε να δώσουμε βοήθεια όμως και στις δύο χώρες ε, το σύστημα επιθεωρητών εργασίας έχει αποδυναμωθεί και αποδιαρθρωθεί και έχουμε διαπιστώσει ότι στην οικοδόμηση διοικητικών μηχανισμών τη στιγμή που έχουν αυτοί ε, αποδυναμωθεί ή δραστικά περιοριστεί είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω με το κατάλογο μου ή αν ε, πρέπει κάπου μόνη να σταματήσω, γιατί φοβούμαι ότι θα σας κουράσω και θα χάσω το κρατήριό μου αν συνεχίσω. Διαφορετικά θα μπορούσα να σας πω για την Ονδούρα και το Ελσαλβαδόρ και μετά να σταματήσω. Ή αλλιώς να θέλετε να, να υποβάλλετε ερωτήσεις. Ναι. Όχι, θα σας κάνουμε ερωτήσεις. Η Άγνες είναι η πρώτη. Ευχαριστώ. Είμαι ευτυχής που έχουμε αυτή την ευκαιρία. Διότι η ερώτησή μου εστιάζεται σε μια από τις χώρες που δεν είναι στον κατάλογό σας, διότι πιστεύω πως κατά κάποιο τρόπο Ίσως ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια και αυτό είναι, αυτή η χώρα είναι το Μπαγκλαντές και επειδή μιλάμε για το Μπαγκλαντές εν γέννη πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να πιέσουμε για την εφαρμογή των προτύπων του Διεθνούς Γραφείου Εργασία. Παίρνοντα αυτό το παράδειγμα του Μπαγκλαντέ, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι σε αυτόν τον κατάλογο, διότι κατά κάποιο τρόπο θεωρήσατε πως ε, έχει γίνει πολύ ισχυρή πρόοδος Ε, και γι' αυτό δεν ε, έχετε καλέσει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να έρθει να απέναντι στην Επιτροπή. Ωστόσο, η χώρα ακόμα ε, αποφελείται από το πρόγραμμα όλα εκτός από όπλα και ειδικά όσον αφορά την εξαγωγή ρουχισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος του Μπαγκλαντές. Το, η χώρα αυτή έχει δεσμευθεί, ωστόσο συνεχίζει συστηματική παραβίαση των ε, βασικών ε, εργατικών δικαιωμάτων και η Κομισιόν ε, επέβαλε δύο προθεσμίες στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πέρυσι, όμως είδα στη δική σας έκθεση προόδου ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος. Οπότε ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ίδια περίπτωση όπως με τη Μιανμάρ ή ίσως άλλους το, άλλες χώρες όπου παράγεται πολύ ρουχισμός. Πρώτον, λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να ξεκινήσει μια επίσημη έρευνα του συστήματος των γενικευμένων προτιμήσεων και δεύτερον, Δεύτερη μου ερώτηση. Από τη δική σας ε, προοπτική για χώρες όπως το Μπαγκλαντές, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε το Βιετνάμ, τη Μιαμάρα, μήπως λοιπόν χρειάζεται πιο δεσμευτική νομοθεσία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, για να εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείε το σεβασμό των εργατικών δικαιωμάτων και εν γέννη θεώρησα και εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, δουλειά που κάνετε στη Γενέβη, αλλά που και που φοβάμαι πως χάνουμε τη μάχη. Πώς μπορούμε λοιπόν να πιέσουμε για καλύτερη εφαρμογή των ε, κύριων συμβάσεων έχετε οποιοδήποτε αίτημα προς τη δική μας κατεύθυνση, ας πούμε για το κοινοβούλιο εδώ ή για το επόμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Βίγκλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ το Κοινοβουλίο για τις ε, πληροφορίες που μας ε, δώσατε γιατί είχατε μια προσέγγιση χώρα ανά χώρα και θα ήμουν ευτυχής να ακούσω μερικά πράγματα παραπάνω για τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Ε, αναφέρατε αυτές τις χώρες, αλλά μόνο σε σχέση με την υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα και άλλες πληροφορίες που θα μπορούσατε να μας δώσετε. Ε, βεβαίως ε, θα υπάρξει και η συνδιάσκεψη Διεθνούς Επιτροπής Μπεωρίου. Επίσης θα ήθελα να, έχω μια, να απαντήσετε μια γενικότερη γενικής φύσεως ερώτηση. Δεν μπορώ να το εκφράσω πολύ κομψά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το διεθνές σύστημα, όχι μόνο το διεθνές σύστημα εμπορίου και ο αλλά όλοι οι διεθνείς οργανισμοί δέχονται την επίθεση πολύ ταραγμένων καιρών. Βλέπουμε ότι στην Ουάσιγκτον υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός και ο ΠΟΕ εφίσταται δρεμίες επιθέσεις και όχι μόνο το Παγκόσμιο Σύστημα Εμπορίου αλλά και άλλες πολυμερείς συμφωνίες. Βλέπουμε την Ουάσιγκτον να αποχωρεί από τη Διεθνή Συμφωνία για το κλίμα ή το πρόγραμμα αφοπλισμού σε σχέση με το Ιράν. Άρα λοιπόν το ερώτημά μου είναι πώς ε, βλέπετε την μελλοντική προοπτική συνεργασίας και πώς βλέπετε το ρόλο του ΠΟΕ ως εταίρου στο Διεθνές Σύστημα Εμπορίου. Γιατί βεβαίως θα πρέπει να επανέλθουμε στις εμπορικές ε, πτυχές που είναι αυτές που μας αφορούν πιο άμεσα. Επίσης θα μου περίεργος να μάθω πώς ε, βλέπετε το μέλλον των πολυμερών συζητήσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί καταρχήν υποστηρίζουμε μεν το πολυμερές εμπορικό σύστημα και έχουμε μια ευαισθησία σχέση με τις εργασιακές ε, πτυχές αυτών των σχέσεων αλλά εν παραλίλω θα πρέπει να προχωρήσουμε και με τις διμερείς μας συμφωνίες. Άρα λοιπόν, πώς βλέπετε τη συνεργασία μας σε αυτό το πλαίσιο, το βαθμό συμπερίληψης των εργασιακών πτυχών στις εμπορικές συμφωνίες, γιατί τελικά αυτό είναι το θέμα που μας αφορά. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Ρένα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε. Δύο χώρες ε, που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερως είναι το Ουσπεκιστάν, όπου υλοποιήθηκε μια συμφωνία με ένα ψήφισμα όσον αφορά το σεβασμό της μη εργασίας των παιδιών και της κατάργησης των, της καταναγκαστικής εργασίας. Ε, Πού βρίσκεται ο ΠΟΕ σε σχέση με τις χώρες αυτές, γιατί Εφόσον συνάψαμε μια συμφωνία, τη συνάψαμε με τον όρο του σεβασμού αυτών των προϋποθέσεων. Το δεύτερο είναι η Κολομβία, επίσης μια χώρα με την οποία έχουμε μια στενή εταιρική σχέση, Κολομβία, Περού και Εκουαδόρ. Ε, με τη νέα πολιτική κατάσταση στην Κολομβία φαίνεται ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο πλαίσιο των συμφωνιών με τον ΜΠΟΕ και των συνδεκάτων και τη συνεργασία με τα συνδικάτα. Οι πολιτικέ τηλεφωνίε ε, αυτή τη βδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ε, κέριο πλήγμα. Ποια είναι λοιπόν η θέση όσον αφορά τι δύο αυτές χώρες. Και τώρα θα ήθελα να πω το εξή ε, το ζήτημα της επικύρωσης των κανόνων του ΠΟΕ αυτό είναι μια πρώτη φάση. Στη συνέχεια είναι και ο σεβασμός αυτών των κανόνων. Ποιος είναι κατά την άποψή σας ε, το σημαντικό εργαλείο που θα πείσει τις επιχειρήσεις και θα τις συμπεριλάβει ε, στην προσπάθεια σεβασμού αυτών των κανόνων. Τι προβλέπετε για τις επιχειρήσεις όσον αφορά το σεβασμό αυτών των κανόνων. Κύριε Σταφίδας. Κύριο Φίσας, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την εκπλήρωση των ε, κανόνων του ΠΟΕ σχέση με την Ιωπανία, θα ήθελα να μάθω αν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σέβονται όλες τις εργασιακές ε, συμβάσεις με τον ΠΟΕ ή αν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή χώρα που δεν δισεύεται πλήρως. Γιατί ε, ας πούμε ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου ε, προσπαθούμε να δώσουμε διδάγματα. Ε, κουνάμε το δάχτυλο και λέμε ότι θα πρέπει να ε, τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις. Πολύ καλή ερώτηση, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ε, ναι, πράγματι είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση και θα συνεχίσω με τη συμφωνία για την, με την Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει έχετε ένα χρονοδιάγραμμα, μια περίοδο προγραμματισμού προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση την οποία περιγράψατε και συμπίπτει με το χρονοδιάγραμμα επικύρωσης της συμφωνίας. Έχει αλλαγή της κατάστασης άμεση επίπτωση στην κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνία. Δεύτερον, αναφέρατε ή αναφέρθηκε προηγουμένως η αναφερθηκε προηγουμενω η κολομβια Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω και το Περού. Γιατί τα πράγματα εκεί δεν αλλάζουν. Το θέμα λοιπόν των εργασιακών συνθήκων στο Περού συνδέονται με τη μετάβαση προκειμένου να δημιουργηθούν ε, διαφορετικές εργασιακές ε, προϋποθέσεις για τους ε, πολίτες αυτής της χώρας. Τρίτον, τύπης, ε, εν γέννη έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια γενικότερη επιδείνωση όσον αφορά το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχει κάποια πρόοδος βεβαίως, αλλά υπάρχει μια μαζική πιστοχώρηση. Πιστεύετε ότι οι βελτιώσεις συνδέονται με την αύξηση της συνδυτότητας, δηλαδή χρειαζόμαστε, από την άλλη χρειαζόμαστε μια, ένα πιο αυστηρό έλεγχο. Ε, τι σκέφτεται η συμπερίληψη δεσμευτικών ρητρών στις συμφωνίες, σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου οι χώρες αυτές να αλλάξουν τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων τους. Γίνεται μια σχετική συζήτηση, γίνεται μια σχετική συζήτηση στον ΠΟΕ ή στο πίπεδο των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την δημιουργία τέτοιου είδους δεσμευτικών προϋποθέσεων. Ευχαριστώ. Η Μαρή Βίνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και κυρία Βάργα. Είπατε ότι θέλετε να ακούσετε τις ε, σκέψεις ε, μας και έχω κάποιες ε, ερωτήσεις. Η Ιαπωνία δεν έχει κυρώσει τις συμβάσεις περί διακριτικής μεταχείρισης ε, και, διακριτική... και καταναγκαστικής εργασίας, ούτε η Σιγκαπούρη, ούτε το Μεξικό. Και λέτε ότι η Ιαπωνία δεν τηρεί και συμβάσεις που έχει υπογράψει, ε, ανεξαρτήτως από όλα αυτά. Πόσο σημαντικό είναι οι βασικές αυτές συμβάσεις να υπογραφούν πριν συμφωνήσει ε, σε μια σύμβαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πόσο επικίνδυνο είναι να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Και να αφαιτώ σε αυτό που είπε και ο κ. Φίσας, ότι το θέμα αφορά και τους τοπικούς αλλά και το τι κάνουμε και εμείς με τα δικαιώματα των ε, συνδικάτων. Μετά, οι μηχανισμοί κυρώσεων, είναι γνωστό βεβαίω ε, το τι συμβαίνει με το Βιετνάμ και η εμπορική συμφωνία μας με αυτήν την χώρα περιέχει κάποια σχετικά κεφάλαια αλλά δεν υπάρχει ένας μηχανισμός κυρώσεων. Στην σύμβαση με το Μεξικό υπάρχουν ε, κάποιες ε, προβλέψεις για την καταβλέψη διαφθοράς. Ωραίο αυτό, αλλά πάλι δεν έχει κάποιο μηχανισμό κυρώσεων. Πώς το βλέπει ο ΑΕΛΟ το θέμα. Ε, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ε, για να έχουμε μια πιο έντονη επιβολή κυρώσεων ή θεωρείτε ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια άλλη προσέγγιση και πώς βλέπετε το θέμα του Βιετνάμ ε, όσον αφορά την καταβλέμηση και της επιρροής της Κίνας και τέλος Θα ήθελα να ακούσω εάν υπάρχει μια πιο θετική άποψη από μέρους σας για το Μεξικό και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Είχα και εγώ μια γενική ερώτηση. Είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γνωρίζω ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μια παρόμοια συζήτηση και στον Καναδά για την επιβολή των σχετικών διατάξεων και από τη σκοπιά του ILO θα ήθελα να ακούσω την δική σας την άποψη για το πώς μπορούμε καλύτερα να επιβάλλουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Η Μάριτα ανέφερε την Κολομβία, θα το έλεγα και εγώ. Οι ΙΠΑ έχουν την συμφωνία για τα παράλληλα ε, εργασιακά δικαιώματα. Εμείς έχουμε τον οδικό χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει κάποιος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα και είναι κάπως ασθενή στο τωρινό πλαίσιο για να αποφύγουμε μια οπισθοχώρηση σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση όσον αφορά τους συνδικαλιστές και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Ένα άλλο παράδειγμα επίσης είναι η Ονδούρα, όπου έχουμε την Συμφωνία της Κεντρικής Αμερικής, έχουμε το κεφάλαιο εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα εργαλεία που έχουμε στην ε, διάθεσή μας για να επιβάλλουμε τα σχετικά κεφάλαια, για να υπάρξει μια πρόοδος, για να βελτιωθεί η ασφάλεια των ακτιβιστών, ε, των συνδικαλιστών και η Αν μου έκλεψε και το θετικό ερώτημα, γιατί πρέπει να είμαστε και θετικοί. Αναρωτιέμαι αν έχει υπάρξει κάποια ένδειξη από τη νέα κυβέρνηση του Μεξικού για το πώς βλέπουν τα εργασιακά δικαιώματα. Επίσης ε, υπάρχει το θέμα του συνδικαλιστή των μεταλλορίχων ε, ο οποίος ε, τώρα ενώ είχε διωχθεί επί σειρά ετών είναι πλέον υπουργό και είναι κάτι το φανταστικό αυτό. Οπότε έχει υπάρξει κάποιο μήνυμα από την κυβέρνηση της ε, χώρας για αυτά τα ζητήματα, για τις βασικές παραβιάσεις εργατικών δικαιωμάτων και για το εργατικό δίκαιο. έχει Σούστερ. Όχι. Μάλιστα. Να πω και εγώ τότε κάποια πράγματα. Το θέμα της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν την Κολομβία και το Περού. Συναντηθήκαμε με την Αμερικανική ομάδα εργασίας και ακόμα και αυτοί μας είπαν ότι δεν υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για να δουν την εφαρμογή. Και ο Καναβάς έχει μια συμφωνία με την Κολομβία, κάπως ε, διαφορετική, αλλά προς την ίδια κατεύθυνση. Και αυτοί επίσης ε, κοιτάνε το ζήτημα της εφαρμογής, αλλά δεν υπάρχει κάποια ενιαία προσέγγιση για έναν μηχανισμό παρακολούθησης ε, της εφαρμογής. Και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του ΑΕΛΟ στο να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους ίσως στην παρακολούθηση της εφαρμογής τέτοιων συμφωνιών. Νομίζω ότι είναι σοβαρό αυτό το πρόβλημα πέρα από την κύρωση των συμφωνιών για να έχουμε έναν κανονικό μηχανισμό παρακολούθησης ε, της εφαρμογής. Και αυτό σχετίζεται και με το θέμα που, ε, που θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην ξεχάσω καμία από τις ερωτήσεις Θα απαντήσω καταρχάς σε κάποιες από τις ερωτήσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένες χώρες ε, για τον Μπαγκλαντές. Οι ερωτήσεις που θίξατε είναι αυτές που πρέπει να θέσει κανείς. Ίσως να σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες για το λόγο που το Μπαγκλαντές δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κατάλογο. Όπως ίσως θυμάστε, το Μπαγκλαντές συζητήθηκε πέρυσι. Δεύτερον, ποιος αποφασίζει ποιες είναι οι 24 χώρες. Οι δύο αντιπρόεδροι της Επιτροπής παίρνουν από κοινού αυτή την απόφαση. Αυτά καταλήγουν σε έναν συναντικό κατάλογο και αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με ένα πρώτο γύρο 40 χωρών και μετά καταλήγουν στις 24. Η επιλογή τους αυτή γίνεται επί τη βάση κάποιων κριτηριών που είναι δημόσια, μεταξύ αυτών σοβαρότητα των θεμάτων, ε, κατά πόσο είναι ε, μόνιμα χαρακτηριστικά, Επίσης εξετάζεται η εξασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στις θεμελιώθεις συμβάσεις και τις κυβερνητικές συμβάσεις και τις ε, τεχνικές. Επίσης προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ισορροπία ανάμεσα στις ε, περιφέρειες, να μην υπερεκπροσωπείται μία περιφέρεια στις συζητήσεις για να αναφέρουμε κάποια κριτήρια. Δεν, είναι όμως ακριβής επιθύμη, οπότε δεν είναι δυνατόν να, τη πληρώσει κανείς όλα τα κριτήρια και να καταλήξει στην τέλεια επιλογή. Υπάρχουν διάφοροι ε, άλλωστε παράγοντες οι οποίοι επίσης ε, λαμβάνονται υπόψη, αλλά το να μην είναι κανείς στον κατάλογο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην λόγω χώρα, γιατί ήταν στη λίστα και δεν είναι πια. Δεν θα πρέπει δηλαδή να θεωρηθεί ότι επειδή δεν είναι στο κατάλογο όλα πάνε καλά. Ρωτάτε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν έχει έρθει ο, ο, κατάλληλη στιγμή για έρευνα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για τα την τήρηση των εργατικών ε, προτύπων και προδιαγραφών. Θα ξέρετε ότι το Γραφείο Εργασίας δεν έχει ε, συγκεκριμένη γνώμη για το κυρώσεις ή την ε, έρευνα. Αυτό είναι απόφαση που πρέπει να λάβουν οι δικοί σας θεσμοί και όπου εμείς δεν έχουμε κάποια επίσημη θέση. Το Μπαγκλαντές είναι αλήθεια ότι όλοι έχουμε την ίδια αίσθηση ανυπομονησίας. Πολλοί χρόνος, πολλή ε, στήριξη, βοήθεια έχει δοθεί, συμβουλές έχουν προσφερθεί, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Μέχρι το Σεπτέμβριο υποτίθεται ότι θα υπάρξει νέα νομική μεταρρύθμιση που θα έχει ολοκληρωθεί. Άρα δεν έχουμε ακόμα ε, συγκεκριμένα στοιχεία. Ίσως ε, το Σεπτέμβριο μπορεί να έχουμε μια νέα <coughs> ρύθμιση, αλλά μπορεί και όχι. Θα πρέπει να το δούμε και να το συζητήσουμε. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Τι μπορεί να κάνει ποιος, ε, με ρωτήσατε. Όσο πιο πολύ ενώνουμε τις δυνάμεις μας και οθούμε προς την ίδια κατεύθυνση, τόσο πιθανότερο είναι ότι θα φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και θα έχουμε κάποιον αντίκτυπο. Όταν κάποια χώρα λαμβάνει μαζικά στήριξη, όπως το Μπαγκλαντές, σε συνεργασία υπάρχουν κάποιες φάσεις όπου η συζήτηση μπορεί να γίνει λίγο πιο δύσκολη, πάντως τα θέματα πρέπει να τεθούν για να έχουμε μια πραγματικά ειλικρινή και έντιμη συζήτηση για το αν και κατά πόσο κινούνται τα πράγματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε πρόσφατη συνδιαλλαγή, ε, μάλλον ε, ε, συζήτηση. Υπήρξε μια ειλικρινή συζήτηση με τον, ε, τους εταίρους από τον Μπαγκλαντές. Εμείς από την ε, πείρα μας στο, στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας θα πρέπει να μένουμε σταθεροί στις αρχές μας, να επαναλαμβάνουμε τα όσα πρέπει να λέμε κάθε φορά ξανά και ξανά κάποιες φορές και με δύσκολες συζητήσεις να μην εγκαταλείπουμε ποτέ την προσπάθεια και ότι τελικά βλέπουμε αποτελέσματα. Ε, υπάρχουν ε, θετικά στοιχεία, γίνονται διάφορες συζητήσεις με την ίδια κυβέρνηση και από διάφορες πλευρές. Γι' αυτό βλέπω ότι έχουμε συμπληρωματικό ρόλο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πιστεύω πως τώρα η κυβέρνηση πήρε το μήνυμα ότι επικρατεί ανυπομονησία και στην Επιτροπή μας ο εκπρόσωπος των εργαζομένων έστειλε σαφές μήνυμα όταν ολοκληρώθηκε η διάσκεψη όπου είπε ακριβώς αυτό ότι δηλαδή θέλουμε να συζητήσει τον Μπαγκλαντές αυτό το θέμα δεν τα κατάφερε εμάς, εμείς ανησυχούμε πολύ εμείς θα παρακολουθούμε και την κατάσταση πολύ στενά και αν δεν υπάρξει πρόοδος μπορεί να προχωρήσουμε σε ε, καταγγελία τύπου άρθρου 26 του χρόνου Υπάρχει αυτό το μήνυμα. Το υπεπτικό σύστημα προσφέρει διάφορους διάβλους για να μπορέσει να καλέσει τις κυβερνήσεις να ε, λογοδοτήσουν σε σχέση με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις και εργοζόμενοι σίγουρα έστειλαν σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνετε αυτό που υποσχεθήκατε. Διότι θα ενεργοποιήσουμε την διαδικασία. Αυτό για τον Μπαγκλαντές. Για την Μιανμάρ και για το Βιετνάμ. Χάνουμε τη μάχη. Όχι. Όχι. Περισσότερο όχι για το Βιετνάμ και λίγο λιγότερο όχι για την ε, Μιανμάρ. Όσον αφορά το Βιετνάμ, πιθανότατα θα γνωρίζετε ότι έχουμε ε, προβεί σε πολύ ε, ε, σοβαρέ συζητήσει με την κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια και θα είμαστε σε μια φάση όπου βλέπουμε την αρχή υποσχόμενων αποτελεσμάτων αυτή της μακρόχρονης συνεργασίας. Έχουν ένα πρόγραμμα για να προχωρήσουν στην επικύρωση των τριών κυρίων συμβάσεων εάν θυμάμαι καλά, 98 σύμβαση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μέχρι το 2019 για την εξάλληψη της καταναγκαστικής εργασίας μέχρι το 2020 και για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε πιθανότατα το, εντός του 2023. Τα μηνύματα είναι όλο ένα και πιο ισχυρά σε σχέση με αυτά τα θετικά βήματα του από πλευράς Βιετνάμ και ξέρω ότι ο πρόεδρός σας θα μεταβεί εκεί σύντομα σε ένα σεμινάριο υψηλό επίπεδο που όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν και εγώ θα είμαι εδώ εκπρόσωπος του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Τώρα, Μιανμάρ. Οι σχέσεις μας με την Μιανμάρ, όπως το συζητούσαμε και χαρακτηρίζονται από ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω. Φαίνεται να είναι δυστυχώς ε, ένας χορός με λάθος βήματα. Η Μιανμάρ ήταν στην κατάλογο ε, φέτος και πιστεύουμε πως η αποστολή επαφής θα βοηθήσει να προχωρήσουμε ε, σε βήματα μεταρρύθμισης και να πιέσουμε για συγκεκριμένες ενέργειες για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με το 87. Νομίζω πως ε, είναι πολύ καλά συντονισμένη η συζήτηση στο ΚΑΣ και τα συμπεράσματα της Επιτροπής σίγουρα θα βοηθήσει το ILO και τον, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε με κοινή ατζέντα για τη Μιαμάρ. Έχουμε ευκαιρίες να διατηρήσουμε την ε, προσήλωσή μας στα θέματα. Τώρα, ε, για το Ουσβεκιστάν, σας πω πού, πού, πού είμαστε. Ε, η πρόοδος ήταν αξιοσημειωτή όσον αφορά την εργασία των παιδιών. Ιδιαίτερα για την παραγωγή και την ε, συγκομιδή Βάμβακος, αλλά και γενικότερα είχαμε συζητήσεις με την κυβέρνηση που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε πριν από λίγα χρόνια. Απλώς ε, αποδοχή της πρακτικής καταναγκαστικής εργασίας ε, και αν το αναγνώρισαν. Έχουν επίσης γίνει συγκεκριμένες ρεύνες που επιτρέπουν τώρα να κάνουμε συζητήσεις πολύ πιο στοχοθετημένες για να εντοπίσουμε συγκεκριμένες δράσεις πολύ συγκεκριμένες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε από κοινού προς πολιτικές που θα, θα περιορίσουν το πρόβλημα της καταναγκαστικής εργασίας, μάλλον της καταναγκαστικής κινητοποίησης για την συλλογή του βάμβακος. Να θυμίσω επίσης ότι η δέσμευση με το Ουσβεκιστάν οδήγησε στην έγκριση της σύμβασης του 87 για την συνδικαλιστική ελευθερία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και φτάσαμε τώρα στο να αναπτύξουμε μια πλήρη συνεργασία για ένα πρόγραμμα που, λέει, που λέγεται αξιοπρεπής εργασία ε, ώστε να έχουμε αναπτύξει ευρύτερη συνεργασία. Ο αρχικό μα εταίρο είναι αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Ε, είναι μια κυβέρνηση προοδευτική ε, που έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις πολλά υποσχόμενες ευρύτερα. Πιστεύω λοιπόν πως το Ουσμπεκιστάν παραμένει και πρέπει να μας χρησιμεύσει σαν παράδειγμα όταν ε, σε κάποιες φάσεις ε, τίνουμε να απελπιζόμαστε ή να προβληματιζόμαστε όταν τα πράγματα αργούν, όμως υπάρχουν αποτελέσματα. Κολομβία. Δύο λόγια για την Κολομβία. Δεν είναι... Ε, όλοι σας ακούσαμε Όλοι μας ακούσαμε, συγγνώμη, τα, τσεκθέσεις για την αύξηση της βίας στην Κολομβία, ιδιαίτερα στον αφορά τους συνδικαλιστές. Πιστεύω ότι αυτή πράγματι είναι μια χώρα όπου ε, κάναμε πράγματα. Ε, βεβαίως ε, δεν έχουμε φτάσει στο τέλος ταξιδιού, ούτε η χώρα έχει ξεπεράσει όλες τις ανταπεξέλθει όλες τις προκλήσεις. Είναι μια χώρα που χρειάζεται υποστήριξη. Ε, είχαμε μια σχετική εμπειρία και ορισμένοι συνάδελφοι μίλησαν πιο λεπτομεριακά σε σχέση με την συνεργασία με την κυβέρνηση Κολομβίας και την Επιτροπή ε, Διευθέτησης ε, Διενέξεων Εργασιακών και ταυτόχρονα εν, εκ με αυτό το οποίο διαβάζετε στον τύπο ε, υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ε, στην Επιτροπή Ελευθεριών και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε διεθνές επίπεδο και να δώσουμε δυνατότητα στην Επιτροπή αυτή να λειτουργεί σωστά εδώ το ILO επικεντρώνει ένα μεγάλο κομμάτι της προσοχής τους προκειμένου να βοηθήσει τη χώρα να επιλύσει τα προβλήματα τοπικά πριν ε, ε, γίνει το πέρασμα στο, στην, ε, στο σύστημα εποπτείας. Προσπαθούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε την Κολονδία σε αυτή την συγκυρία που βρήθη προκλήσεων. Το Μεξικό. Ακούσαμε τίποτα από την ε, πρόσφατα εκλεγήσα κυβέρνηση. Νομίζω ίσως ότι είναι πολύ νωρίς. Αναμένω η νέα κυβέρνηση να οικοδομήσει στην, στο έργο που επιτελέσαμε από κοινού με την προηγούμενη κυβέρνηση Άλλο όπως σας είπα, είναι πολύ νωρίς ε, για να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκα σε όλες τις ε, χώρες που ε, που αναφέρατε. Τώρα, όσον αφορά τη, γενική έννοια μιας παγκόσμια επιδείνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, θα ήθελα να πω ότι πάντοτε είμαι κάπως προσεκτική με αυτές τις ε, γενικεύσεις που βεβαίως έχουν σωστές ε, εφόσον στηριχθούμε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο τεκμηριώνει αυτήν την υπόθεση αλλά μπορούμε να βρούμε ένα ακριβώς αντίθετο παράδειγμα. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να προσεγγίσουμε τη συζήτηση αυτή, την προβληματική αυτή με σύνεση και ενδεχομένως να κάνουμε περισσότερες ε, διαφοροποίησεις σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα σε συνάρτηση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, αν δούμε τα δικαιώματα των παιδιών, δεν θεωρώ ότι στέκει η θέση μιας ε, γενικής επιδίνωσης. Θεωρώ ότι εδώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την ε, μείωση της παιδικής εργασίας. Βεβαίως δεν έχει εξαλειφθεί. Υπάρχουν 600 εκατομμύρια παιδιά τα οποία εργάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός. Παρ' όλα αυτά έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο και η αριθμή αυτή ήταν πολύ ψηλότερη μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Απομένουν ε, προκλήσεις ε, βεβαίως και πιστεύω ότι η παιδική εργασία ασφαλώς είναι ένα καλό παράδειγμα για το εξή. Εάν η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιήσει τις δυνάμεις της, όπως συνέβη με το θέμα αυτό, σε σχέση με τις ε, χειρότερες ε, μορφές της παιδικής εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα να σημειωθεί κάποια πρόοδος τώρα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση κατά πόσο έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των όσων έχουμε πετύχει. Αυτή είναι μία πτυχή βεβαίως που αφορά το γενικότερο περιβάλλον που πρέπει να έχουμε κατά νου. Και αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού είναι να αποφύγουμε οι συνταγές ε, προώθησης οικονομικής μεγέθυνσης σε μια δύσκολη συγκυρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης ε, το πολυμερές ε, μοντέλο το οποίο αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί από πεπαλαιωμένες συνταγές και φόρμουλες οι οποίες ξανάρχονται στο προσκήνιο. Νομίζω ότι η απειλή, ή συγγνώμη, η πρόκληση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το να διατηρήσουμε ζωντανή, ε, μάλλον, την προσοχή όλων μας σε μία ίση ανάπτυξη, έστω και σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκύρια. Κανείς θα μπορούσε να σκεφτεί γρήγορο, γρήγορα κέρδη λαμβάνοντας σκληρές οικονομικές αποφάσεις για ορισμένε χώρες και για να παρέλθω στη Μολδαβία, την Ουκρανία η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ε, ε, και στη συνέχεια ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων που που ανακύπτουν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι βασικοί οργανισμοί εργασίας θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να επαγρυπνήσουν για την ε, ε, κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί Εάν επιστοχωρήσουμε σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, ε, τα κέρδη που θα αποκομίσουμε θα είναι πενιχρά. Τώρα, σε αυτές τις ε, ταραχώδεις ε, εποχές για το πολυμερές σύστημα, προφανώς δεν έχουμε ανοσία και στον ILO έναντι της περιραίωσης αυτής της ατμόσφαιρας. Ε, Παρ' όλα αυτά πρόσφατα ε, στη συνδιάσκεψη του ΑΕΛΟ ακούσαμε πολλούς να υποστηρίζουν το πολυμερές μοντέλο εντός του ILO. Δεν υπήρξαν ενδείξεις δηλαδή που να μας λένε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες θέτουν ένα αμφιβόλο το σύστημα του πολυμερού συστήματος. Και τέθηκε μία ερώτηση σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει η μετατόπιση από το πολυμερές σύστημα προς ε, διμερείς ε, συμφωνίες. Αυτή είναι μια ερώτηση που το ΑΕΛΟ δεν μπορεί να έχει μια επίσημη τοποθέτηση. Αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ένα ισχυρό κεφάλαιο για τα εργασικά δικαιώματα. Εάν αποδυναμωθεί το πολυμερές ε, σύστημα, η σύναψη ε, διμερών συμφωνιών θα δυσχερανθεί πολύ και με όρους των κεφαλαίων περί εργασίας, σίγουρα το ILO ε, προσπαθεί να διατηρήσει το, πολυμερές, το μοντέλο των πολυμερών σχέσεων. Θέστε πολλά ερωτήματα. Εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών και ενδεδειγμένος μηχανισμός ε, παρακολούθησης, εποπτείας, ε, θα πρέπει να υπάρξει μια... Ε, έχει γίνει, συγγνώμη, μια επισκόπηση της, ε, των εξελίξεων, της προόδου της κάθε χώρας και υπήρξαν κάποια εντυπωσιακά αποτελέσματα. Υπάρχουν κάποια δεχνή φόρα τα οποία συζητούν τα θέματα αυτά και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς ε, να συνεχίζει να ασκεί πίεση ως προς τα θέματα αυτά. Βεβαίως αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν πιστεύω ότι η επιτήρηση η ίδια, η εποπτεία η ίδια ε, σφαίρει αποτελέσματα. Η ενεργός ε, δράση μέσω της συνεργασίας με τις χώρες μέλη είναι πιο πρόσφορη και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να πάνε χέρι-χέρι. Και Ενδεχομένω θα πρέπει να υπάρξει μια εκ παρακολούθηση αυτών των μορφών συνεργασία, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κινούμεθα προς ε, ένα πιο στέρεο σύστημα, πιο ρωμαλαίο σύστημα εποπτείας. Πολλοί από εσά ε, ανέφεραν το ζήτημα της συμμόρφωσης. Ποιος συμμορφώνονται πλήρως. Συμμορφώνονται πλήρως οι ευρωπαϊκές ε, χώρες με αυτούς τους ε, κανόνες. Ασφαλώς όχι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε είναι ένας μηχανισμός τακτικής ε, παρακολούθησης των θεμάτων των πτυχών ε, συμμόρφωσης προκειμένου να υποστηριχθούν οι χώρες ως προς την τήρηση των δεσμεύσεών τους. Από κοινού με το Φόρουμ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιχειρήσεις. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε δράσεις μεταξύ κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ευρύτερους, ευρύτερες συμμαχίες και με τις επιχειρήσεις και να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις πιο υπεύθυνε και διατεθειμένες να συμπεριλάβουν όλα αυτά τα θέματα στις δικές τους προσπάθειες Ε, γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας ε, κίνδυνος μη συμμόρφωσης και θα πρέπει εδώ στη βάση αυτή να οικοδομήσουμε. Thanks Ευχαριστούμε. πολύ. Ναι, ναι. Σωστά απαιτείται πράγματι εμπλοκή σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, η Κομισιόν ίσως έχει κάτι να μας πει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εξπακούεται ότι η σωστή εφαρμογή των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική και αναγνωρίζουμε οπωσδήποτε τον ρόλο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Απασχόλησης έχει πολύ καλή συνεργασία με τον και θεωρούμε ότι ο πολυμερής αυτός οργανισμός παίζει κέριο ρόλο στην εμπορική μας ε, πολιτική και βεβαίως ε, παρακολουθούμε το πώς εντείνεται ο ρόλος του. Βλέπουμε ότι είχαμε συγκεκριμένο αντίκτυπο από τις ε, θεμελιώδεις συμβάσεις ε, του ILO και δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω εγώ πως είχαμε μονομερείς ε, προτιμήσεις υπό το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων. στο σύστημα Everything But Arms, τα πάντα εκτός από όπλα, όπου έπαιξε έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η προσχώρηση των κρατών στις συμβάσεις ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την ε, σύναψη συμβάσεων. Και βέβαια υπάρχει το θέμα της σωστής ε, εφαρμογής ειδικά των κεφαλαίων για τα εργασιακά και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και βεβαίως έχουμε τα θέματα της καταναγκαστικής εργασίας. Έχουμε και κλαδικούς φακέλους, ε, παραδείγματος χάρη φαντουργία, τρόφιμα με το Μπαγκλαντές. Και εδώ έχουμε ακριβώς και την τέταρτη συνεδρίαση του Συμφώνου Αηφορίας ε, πριν από 15 μέρες και στείλαμε έντονα μηνύματα στις αρχές των Μπαγκλαντές ε, από όλους τους μας και από τον Επίτροπο Εμπορίου που επέμεινε στο ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος ειδικά στα ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων ε, στις ε, προτιμήσεις για τα πάντα εκτός από όπλα. Και ακριβώς ακούσαμε από τους συνομιλητές μας ότι σκοπεύουν ε, τον Ιούλιο να προτείνουν ε, ένα νομοθετικό πακέτο αφορά <coughs> τα εργασιακά και τις ειδικέ οικονομικές ε, ζώνες και είχαμε ακριβώς και μια αποστολή αυτόν τον μήνα στην ΕΝΤΑΚΑ για αυτό το ζήτημα. Και ακριβώ ε, θα δούμε και τον Υπουργό Εμπορίου για αυτό το ζήτημα. Επιπλέον θα πάμε και τον Σεπτέμβριο στην ΝΤΑΚΑ για να δούμε ακριβώς την πρόοδο που μας υποσχέθηκαν στην ε, συνεδρίαση που έγινε στις Βρυξέλλες. Σε γενικές γραμμές λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε επίσης ε, πολλές επαφές ε, με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για την κύρωση των συμβάσεων και θεωρώ ότι έχουμε αργά αλλά σταθερά αποτελέσματα. Συμπερασματικά λοιπόν θα ήθελα να πω ότι η Κομισιόν στηρίζει πλήρως ε, το πολυμερές ε, σύστημα και ελπίζω για το ότι αποτελεί μια βασική ε, πηγή έμπνευσης για την πολιτική μας για το εμπόριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Τελειώσαμε με το σημείο 14. Καλή τύχη σας εύχομαι, κυρία Βάργα. Το επόμενο θέμα, το 15, είναι και κλεισμένων των θυρών. Θα σταματήσει και η μετάδοση στο διαδίκτυο. Ε, παρακαλώ όσοι δεν έχουν εργασία να φύγουν από την αίθουσα. Διέρμα λίγων λεπτών.